σημείο είναι η έκθεση του κυρίου Φλέκενστάιν για την πρόσβαση στην αγορά λιμενικών υπηρεσιών και χρηματοοικονομικών και τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων. Συγγνώμη. Ο κύριος ε, Φλέκενστάιν προέρχεται από μια πόλη λιμάνι. Του δίνω λοιπόν αμέσως το λόγο. Κύριε Φλέκενστάιν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, από την αρχή της συζήτησης για το πακέτο λιμένων 1 πριν από 15 χρόνια ε, κατ' ε, δεν υπήρξε δικαιολογημένα πλειοψηφία στο σώμα. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι το, η σημερινή πρόταση είναι βελτιωμένη και θα εγκριθεί γιατί διαφοροποιείται ξεκάθαρα από τις ε, προηγούμενες μια έγκριση και μια εντολή διαπραγμάτευση στο Συμβούλιο είναι εφικτές γιατί η πρόταση δεν ε, δεν μάλλον εκμεταλλεύεται την επιθυμία αύξησης της ανταγωνιστικότητας. Στο επίκεντρο δεν βρίσκεται το άνοιγμα των αγορών, αλλά η καλύτερη οργάνωση των λιμένων μάλιστα με έναν περιορισμό του αριθμού των παρόχων εφόσον κάτι τέτοιο μοιάζει αναγκαίο. Στη σημερινή πρόταση προ... παρόλα αυτά προβλέπεται αύξηση της ανταγωνιστικότητας, μεγαλύτερη διαφάνεια, καλύτερη ενημέρωση των χρηστών και σοβαρή αλλά μη γραφειοκρατική εποπτεία. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας ε, συνεπάγεται ότι υπάρχουν καλές, ε, σωστές ε, θέσεις εργασίες στους λιμένες. Και γνωρίζω ότι με τον κανονισμό τα ζητήματα αυτά δεν μπορούν να ρυθμιστούν, αλλά μία αποτελούν μια επισήμανση για εκείνους που θα μπορούσαν να τα ρυθμίσουν. Αυτό αφορά την καλύτερη εκπαίδευση και κατάρτιση καθώς και εργασιακά μοντέλα τα οποία θα μπορούσαν να εξελιχθούν για να δημιουργήσουν ε, καλύτερες ε, θέσεις εργασίας. Η σημερινή λύση είναι δυνατή γιατί η Επίτροπος Πούλτς ε, σε αντίθεση με τον προκάτοχό της πραγματικά επέλεξε μια συνεργασία ε, με το, με το σώμα ε, και μια ευρεία συζήτηση στην οποία συμμετείχαν πολλοί ενδιαφερόμενοι. Ε, για παράδειγμα, παρόλα αυτά υπήρξαν προβλήματα. Για παράδειγμα, οι Βρετανοί θεωρούσαν ότι δεν αφορά αυτούς ε, το θέμα των, λιμών, των λιμένων. Ε, επίσης, οι Πολωνοί δεν ήταν διατεθειμένοι να το συζητήσουν γιατί δεν ήθελαν να δεχτούν το θέμα της διαφάνειας. Και βεβαίως οι Ευρωπαίοι δεν ήταν ενθουσιασμένοι ε, γιατί το όραμά τους ε, Φιλιππινέζοι ναυτικοί να εκφορτώνουν στους ευρωπαϊκούς ε, λιμένες θα φτάσει σε ένα τέλος. Θα υπάρξει ωστόσο μία ικανοποιητική έκβαση μόνο εφόσον το Συμβούλιο συνεργαστεί με την Επιτροπή όσον αφορά το ζήτημα των ε, συλλογικών ε, ε, των εξαιρέσεων για τις κρατικές ενισχύσεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Ισκιώδης για την εξαίρετη συνεργασία, επίσης την Επίτροπο γιατί επέλεξε την οδό του πραγματισμού και όλους τους ε, ενδιαφερόμενους να, θα ήθελα επίσης να τους ευχαριστήσω, συμμετείχαν στις διαβουλεύσεις γιατί πραγματικά έδειξαν την ε, διάθεση να καταλήξουμε σε ένα απτό αποτέλεσμα. Πραγματικά πρόκειται για ένα καλό συμβασμό και θα ήθελα να σας παρακαλέσω να τον εγκρίνετε αύριο. Η κυρία Μπούλτς έχει το λόγο εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, η Επιτροπή καλωσορίζει την έκθεση που θα συζητηθεί απόψε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Φλέκενστάιν ειλικρινά για τη σημαντική εργασία, ιδιαίτερα εκείνη που προσβλέπει προς το μέλλον. Να ευχαριστήσω και την Επιτροπή Μεταφορών και τους Σκιώδης για την ε, πολύ καλή έκθεση ο κανονισμός για τις λιμενικές υπηρεσίες έχει μεγάλη σημασία για την προώθηση του επενδυτικού τομέα. Ξέρετε το ζωτικό ρόλο των λιμένων για το σύστημα μεταφορών και την οικονομία. Είναι οι πύλες μας προς τον κόσμο. Δημιουργούν απασχόληση και εμπόρια και επίσης ε, θα πρέπει ε, να προωθήσουμε τα έργα αυτά μέσα στα πλαίσια της απομάκρυνσης από τη χρήση του άνθρακα. Όλα αυτά θα πρέπει να ενισχυθούν και γι' αυτό θεωρούμε ότι είναι και ένα από τα βασικά μας χαρτοφυλάκια και προτεραιότητες για το 2016. Επίσης θα γίνει σωστή χρήση των κονδυλίων και θα θέλαμε οι λιμένες να έχουν ίση πρόσβαση στο εμπόριο, να υπάρχει χρηματοδοτική διαφάνεια και να μην υπάρχει προτιμησιακή μεταχείριση. Έτσι θα μπορέσουμε να ε, απλουστεύσουμε και τους κανόνες για την κρατική ενίσχυση. Θα πρέπει να υπάρχουν εξαιρέσεις επενδύσεων, ιδιαίτερα για ορισμένους λιμένες όπου ε, υπάρχει κρατική ενίσχυση, έτσι ώστε να υπάρχει ίση πρόσβαση. Ένα πρώτο προσχέδιο δημοσιεύθηκε σήμερα και σήμερα άρχισε και η δημόσια διαβούλευση. Ο κανονισμός για τις υπηρεσίες λιμένων θα αποτελέσει ένα βασικό input με τη δική σας υποστήριξη. Ο κανονισμός αυτός θα δώσει διαφάνεια και στη διαδικασία δημοπράτησης έτσι ώστε να μην υπάρχει ασάφεια όπου δεν αποφασίζεται η πολιτική από τον νομοθέτη αλλά αναπερίπτωση και από το ΔΕΚ ε, δυνάμει των συνθήκων. Η έγκριση του κανονισμού σημαίνει μεγαλύτερη νομική διαφάνεια και σταθερότητα και για τους επενδυτές και για τους εργαζόμενους. Ο κανονισμός είναι σημαντικός και για την απομάκρυνση από τη χρήση άνθρακα γιατί έχουμε δεσμευτεί γι' αυτό με βάση το COP21. Έτσι η χρήση λιμένων θα γίνει πιο δελεαστική για να αποσυμφορηθούν και οι οδικές μεταφορές. Θα πρέπει να υπάρχει διαφοροποίηση των θαλασσίων οδών και να προωθήσουμε και την αυσιπλοεία μικρών αποστάσεων. Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, η έκθεση υποστηρίχθηκε από την Επιτροπή Μεταφορών. Όλοι οι βασικοί οργανισμοί την υποστηρίζουν. Τα συνδικάτα, οι λιμενικές αρχές, η τερματική σταθμή και οι πάροχοι. Υποστηρίζουμε τον κοινωνικό διάλογο καθώς και την καλύτερη κατάρτιση και ασφάλεια για τους εργαζόμενους. Θα ήθελα να τονίσω ότι ο κανονισμός δεν επιβάλλει ένα κοινό μέτρο για όλους. Ξέρουμε ότι κάθε λιμάνι στην Ευρώπη είναι διαφορετικό και αυτό το σέβεται το προσχέδιο και συμβαδίζει και με την χρήση των ιδιωτικών λιμένων. Δεν επιβάλλει σχήματα. Αύριο θα αρχίσουν οι τριμερείς διάλογοι και έχουν μεγάλη σημασία για την προώθηση αυτού του νομοθετήματος. Το Συμβούλιο ήδη ενέκρινε μια γενική προσέγγιση το 2014. Αυτό ήταν μία από τις μεγάλες επιτυχίες της Ιταλικής Προεδρίας. Θα πρέπει το Κοινοβούλιο να αρχίσει τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο για να λήξει το ζήτημα αυτό. Η Ολλανδική Προεδρία θα ήθελε ήδη πριν από το καλοκαίρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες. Σας καλώ όλους να μην χάσουμε αυτή την ευκαιρία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα θα μιλήσουμε εκ μέρους των πολιτικών ομάδων οι αγορητές. Εκ μέρους του ΕΛΚ καταρχήν η κυρία Βόζεμπερκ Βριονίδη. Ενάμιση λεπτό έχετε στην διάθεσή σας. Κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα λιμάνια αποτελούν αδιαμφισβήτητα ένα από τους σημαντικότερους μοχλούς οικονομικής ανάπτυξης, αλλά και πηγή ευημερίας για τα κράτη-μέλη και την Ευρώπη. Δεν είναι τυχαίο ότι το 75% του εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και το 38% του ενδοκινοτικού εμπορίου διεξάγεται δια θαλάσσης, γεγονός που υποδηλώνει τη σπουδαιότητα του τομέα για το λόγο αυτό ο κανονισμός που θα ψηφίσουμε στην ολομέλεια αποσκοπεί στην ενίσχυση της απόδοσης των ευρωπαϊκών λιμένων και τη βελτίωση της συνολικής ποιότητας των λιμενικών υπηρεσιών με στόχο τον εξυγχρονισμό τους. επίσης δημιουργεί συνθήκες δικαιότερου ανταγωνισμού μειώνει τις νομικές ασάφειες ενδυναμώνει τη διαφάνεια και την καλύτερη κατανομή των δημοσίων πόρων. μόνο η δημιουργία σταθερού νομικού περιβάλλοντος που διέπεται από δίκαιους όρους ανταγωνισμού και συγκεκριμένους κανόνες διαφάνειας διαφάνειας μπορεί να προσελκύσει επενδύσεις στα λιμάνια συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της οικονομίας της ευρωπαϊκής ένωσης ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής κρίσης. παράλληλα η νέα νομοθεσία δίνει στα λιμάνια μεγαλύτερη αυτονομία σχετικά με τον καθορισμό των λιμενικών τελών το γεγονός αυτό ενισχύει τον ανταγωνισμό τόσο μεταξύ των ευρωπαϊκών λιμένων όσο και μεταξύ των λιμένων της ευρωπαϊκής ένωσης με τρίτες χώρες. επιπλέον προβλέπει μια σειρά ευνοϊκών διατάξεων για τα μικρά λιμάνια ώστε να αποφευχθεί η δυσανάλογη διοικητική επιβάρυνση και τα πρόσθετα τέλη και τα κόστη. Η Ευρώπη έχει ανάγκη από τέτοιες νομοθετικές πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν τα κοινά συμφέροντα μεταξύ των κρατών μελών και τονώνουν την ανιαία εσωτερική αγορά. Σα ευχαριστώ πολύ. Uh, uh, Έχετε μπλε κάρτα από την κυρία Γκραπινή. Yes. Okay. <coughs> Κυρία Γκραπινή, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, και εγώ εκτιμώ ότι η έκθεση είναι πολύ σημαντική, όπως μας είπε και η Επίτροπος. Θα ήθελα να σας απευθύνω μία ερώτηση. Η διαφορά μεταξύ αυτού που προτείνει η Επιτροπή και των εισηγητών σχετίζεται με τους δασμούς, με τα τέλη που θα επιβληθούν στους λιμένες. Θεωρείτε ότι θα ήταν σκόπιμο να υπάρξει μία επιτροπή ε, διαχείρισης των τελών ή αυτά να τα ορίζουν οι ίδιοι λιμένες. ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. θα σας πω ότι στο κείμενό μας είναι απόλυτα ισορροπημένο ακριβώς και στον τομέα τον οποίο θίξατε διότι προβλέπει και μια δίκαιη κατανομή των τελών και, του κόστους και για τα μικρότερα λιμάνια που μέχρι στιγμής είχαν μια επιβάρυνση. Στην ερώτησή σας απαντώ ότι διαβλέπει και αυτή την παράμετρο το κείμενο ολοκληρωμένα μάλιστα με ισορροπημένες τροπολογίες που ε, έγιναν κατόπιν πολλών συζητήσεων μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. On behalf SND Group, uh, Deputy... Ευχαριστώ. Εκ μέρου ε, των Σοσιαλιστών, η κυρία Άντερσον για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν πάνω από 300 ευρωπαϊκά λιμάνια στο ευρωπαϊκό δίκτυο και πάνω από 3 εκατομμύρια θέσεις εργασίας εξαρτώνται από τον λιμενικό κλάδο άμεσα ή έμεσα. Και αν δούμε την ποικιλομορφία στη διαχείριση των ευρωπαϊκών ε, λιμάνων, ε, λιμένων θα έπρεπε να ρυθμίσουμε τον κλάδο αυτό με τη μεγαλύτερη προσοχή. Ε, ε ορισμένοι αντιτίθεται στα ισορροπημένα μέτρα εδώ που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αύξηση της ασφαλείας, στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και να παράσχουν ένα ασφαλές πλαίσιο για επενδύσεις. Ωστόσο το πρόβλημα είναι ότι παρά τις προσπάθειες του εισηγητού η πρόταση αυτή δεν επιτυγχάνει τους στόχους που ανέφερα. Υπάρχουν κάποιες προβλέψεις σχέση με την κατάρτιση και την ενθάρρυνση των καλών ε, πρακτικών όσον αφορά τη δημοπράτηση, αλλά όλα αυτά δεν αρκούν. Το σχέδιο κανονισμού είναι ένα παράδειγμα πραγματικά θεαματικών, ε, θεαματικής υποκρισίας διπλών κανόνων και γιατί εξακολουθεί να υπάρχει ένα διοικητικό άχθος για τους ε, λιμένες και δεν υπάρχει καμία σαφήνεια εάν διαβάσει κανείς το κείμενο. Κανείς ε, έχει πολλά ερωτήματα ε, και υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα όσον αφορά την χρέωση των τελών πολλά σημαντικά προβλήματα δεν καλύπτονται από το κείμενο και δεν υπάρχει μια ενημέρωση όσον αφορά τη μελέτη αντιχτύπου και όσον αφορά μια ενδεχόμενη συμφωνία θα έπρεπε τα στοιχεία αυτά για τις μελέτες αντικτύπου να είναι εντελώς επικαιροποιημένα. Εμείς ε, θέλουμε να υπάρχει κάτι το οποίο βελτιώνει τα δικαιώματα των εργαζόμενων. Και πραγματικά αυτό απουσιάζει εδώ. Οι λιμένες ε, ε, οι λιμενικοί φορείς επίσης δεν θα διαβολευθούν με εμπειρογνώμονες του περιβάλλοντος. Με άλλα λόγια θα σας παρακαλούσα να απορρίψετε την πρόταση της Επιτροπής. Ευχαριστούμε πολύ. Δέχεστε μια μπλε κάρτα Ευχαριστώ πολύ, κυρία Άντερσεν. Αναφέρατε τις αμφιβολίες όσον αφορά κοινωνικά θέματα δεν είστε ικανοποιημένοι για τα κοινωνικά δικαιώματα, αλλά ποια είναι η άποψή σας για την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία όσον αφορά αυτή την πρόταση κανονισμού. Ευχαριστώ πολύ. Όσον αφορά το κοινωνικό στοιχείο, πιστεύω ότι θα μπορούσαν να γίνουν πολύ περισσότερα πράγματα στα διάφορα επιμέρου άρθρα για να, ε, για να ενισχυθεί η αξία του κοινωνικού διαλόγου. Γιατί ε, παρόλο που βεβαίως ε, τα πράγματα θα μπορούσαν να ήταν ε, χειρότερα, παρόλα αυτά δεν είμαι απολύτως ικανοποιημένη εδώ. Και αν δείτε τις προηγούμενες θέσεις εν σχέση με το τι ήθελαν οι διάφορες πλευρές του κοινωνικού διαλογού, πραγματικά δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι θα είναι ικανοποιημένοι. Όσον αφορά για την ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία, βεβαίως γίνεται λόγος για τα προβλήματα και αυτό αυξάνει τη συνειδητότητα, αλλά δεν επαρκή. Ευχαριστούμε πολύ. Για δύο λεπτά κυρία... ο κύριος Βαν Ντάλεν. Κύριε Πρόεδρε, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Φλίκενστάιν που τόλμησε με ρεαλισμό να παρουσιάσει το θέμα αυτό και το ΕΛΚΑ και η ECR νομίζω επικρότησαν το έργο αυτό θα ήθελα να αναφερθώ σε ορισμένα σημεία μείωση της γραφειοκρατίας, λιγότερος διοικητικός φόρτος. Αρχικά υπήρχαν πάρα πολλές διατάξεις για κοινωνικά θέματα, υποχρεώσεις για κατάρτιση, για δεξιότητες, για προσόντα, αλλά πολλές υποδομές λιμενικές δεν μπορούν να προσφέρουν τέτοια κατάρτιση και γι' αυτό ευτυχώς καταργήθηκαν αυτές οι διατάξεις. Δεν μιλάμε πια για υποχρεωτική πρόσβαση στην αγορά. Επανερχόμεθα στην κατάσταση που υπάρχει στα κράτη-μέλη και στις περιφέρειες. Τα ίδια τα λιμάνια θα οργανωθούν μόνα τους. Στο Ρότερνταμ η κατάσταση είναι διαφορετική από ό,τι στο Βίγκο, παραδείγματο χάρη. Η επικουρικότητα και η κυριαρχία βρίσκουν εδώ την πλήρη έκφρασή τους. Επίσης προβλέφθηκε μια εξαίρεση για τα ιδιωτικά λιμάνια, τα βρετανικά, τα οποία μπορούν τώρα από μόνα τους να προβλέψουν ειδικέ ρυθμίσεις, όπω παραδείγματο χάρη ε, για τα μέτρα και ε, τα βάρη των ε, πλοίων, για την ρημούλκηση, για τους πιλότους, για τον ελιμενισμό. Ορισμένοι θέλουν να μην υπάρξουν αυτές οι διατάξεις. Αυτό είναι ανόητο διότι η κυρία Βεστέρ της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού θα λάβει διατάξεις και μέτρα τα οποία θα ισχύουν άμεσα για τους λιμένες και θα ανοίξουμε το κουτί της Πανδώρας με τον τρόπο αυτό. Ε, θα, θα ήταν λογικό και στη δική μου την ομάδα. Ξέρω ότι όλοι δεν συμφωνούν. Καλό όλους να υποστηρίξουν αυτή την πρόταση. Εκ μέρους του Άλντε, η κυρία Γκεζίνε Μάισνερ. Ευχαριστώ πολύ, ε, Επίτροπε. Οι λιμένες ε, στην Ευρώπη διαφέρουν μεταξύ τους. Αυτό το διαπιστώσαμε και είναι πολύ δύσκολο να έχουμε ένα κοινό πακέτο για τους λιμένες. Αυτή είναι η τρίτη προσπάθεια και ελπίζω αυτή τη φορά να πετύχει. Ίσως ε, είναι ωραίο που μιλάω μετά από τα, άλλε άλλες πολιτικές ομάδες γιατί βλέπουμε πόσες ε, αποκλήσεις υπάρχουν σε διάφορες απόψεις. Οι σοσιαλιστές είπαν ότι δεν λήφθησαν υπόψη τα κοινωνικά δικαιώματα. Ε, και όλα αυτά ε, δείχνουν ότι πραγματικά ότι ο εισηγητής πέτυχε έναν καλό συμβιβασμό. Βεβαίως δεν είναι δυνατόν να κανοποιηθούν κατά 100% όλα τα αιτήματα. Ε, εμείς, ε, για παράδειγμα, θέλαμε να εξαιρεθούν πολύ περισσότερες ε, υπηρεσίες και να υπάρξουν συγκεκριμένε ρήτρε. Παρ' όλα αυτά θεωρούμε ότι είναι ένας συμβιβασμός ο οποίος είναι βατός για να χωρίσουμε και κατά την άποψή μου εδώ υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό και το οποίο φάνηκε και στις ανακοινώσεις τύπου και το οποίο ικανοποιεί τόσο τα συνδικάτα όσο και τις, ε, τους παρόχους λιμενικών υπηρεσιών. Γι' αυτό παρακαλούμε να εγκριθεί η πρόταση κανονισμού γιατί είναι πολύ σημαντική η θέση των ε, λιμένων. Γιατί εδώ έχουμε μια σχετική διαφάνεια για τις χρηματοοικονομικές ε, ροές, ε, πολύ καλές συνθήκες για τους εργαζόμενους, αλλά και κίνητρα για επενδύσεις. Όλα αυτά εξασφαλίζονται από την πρόταση κανονισμού και γνωρίζω ότι ήταν πολύ δύσκολο, γιατί η πρόταση της Επιτροπής και αυτό το οποίο αρχικά ήθελε ο εισηγητής, πραγματικά δεν μπορούσαν να συνδυαστούν. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε μια μεσαία άποψη ε, και πραγματικά πολλά στοιχεία έχουν συμπεριληφθεί. Ε, τα πάντα δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν. Θεωρώ ότι θα πρέπει να εγκριθεί η πρόταση κανονισμού υπέρ των λιμένων και υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, ο κύριος Κούλογλου έχει το λόγο. Είναι καλό ότι κατορθώσαμε να θέσουμε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο λειτουργίας το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού περιορίστηκε στην οργάνωση των λιμένων και τη διαφάνεια των οικονομικών συναλλαγών. δεν υπάρχουν ρυθμίσεις σχετικές με την απορρίθμιση των εργασιακών σχέσεων και το ανεξέλεγκτο άνοιγμα στις αγορές. πολλοί εμπλεκόμενοι φορείς και τα περισσότερα συνδικάτα υποστήριξαν τη δουλειά μας. κατορθώσαμε το αποτέλεσμα να απέχει από τους αρχικούς στόχους της επιτροπής σε αυτή τη βάση η προσδιαπραγμάτευση με το συμβούλιο πρόταση παρέχει μια καλή προστασία για τους εργαζόμενους στα ζητήματα ασφάλειας και υγείας ενισχύει το δικαίωμα στην εκπαίδευση και κατάρτιση και θα λειτουργήσει σαν ανάχωμα μπροστά σε παραπέρα επιθέσεις ενάντια στις συνθήκες εργασίας. προβλέπει την περιβαλλοντική βιωσιμότητα των λιμενικών υπηρεσιών και όλα αυτά σε συνθήκες διαφάνειας θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τη δουλειά του. σας προτρέπω να ψηφίσετε υπέρ των συμβιβαστικών τροπολογιών που υιοθετήθηκαν σε μπλοκ και να δώσουμε στον κύριο φλέγκενστάιν την εντολή για την έναρξη των διαπραγματεύσεων με το συμβούλιο και την επιτροπή. τώρα τα κράτη μέλη και οι κυβερνήσεις πρέπει να αποδείξουν την ετοιμότητά τους για ισχυρές δεσμεύσεις ενάντια στο κοινωνικό ντάμπινγκ και υπέρ της προάσπισης των ασφαλών εργασιακών συνδικών στα λιμάνια. Ευχαριστώ. Δέχεστε μπλε κάρτα από την κυρία Άντερσον. Um, Ευχαριστώ. Καταλαβαίνω τα όσα είπατε σε σχέση με την ε, πλήρη απελευθέρωση που δεν περιλαμβάνεται σε αυτό το μήνυμα. Παρ' όλα αυτά ε, υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες για τους, ε, για τους διαχειριστικούς φορείς σε σχέση με τους παρόχους λιμενικών υπηρεσιών. Αυτό είναι που σας ενδιαφέρει. δεν ξέρω, ίσως όμως ένα μέτρο περί διαφάνειας στην περίπτωση αυτή θα ήταν παραπλανητικό. Πάρτο, πάρτο. Ε, ε, του Κοινοβουλίου. Πιστεύω ότι υπάρχουν καλοί και κακοί συμβιβασμοί και εδώ έχουμε να κάνουμε με έναν ε, καλό αξιοπρεπή συμβιβασμό που προασπίζει τα βασικά δικαιώματα. Ευχαριστώ. Εκ μέρους των Πρασίνων, ο κύριος Κιφτέιλ. Ευχαριστώ. Μετά από δύο θεαματικές προσπάθειες απελευθέρωσης των λιμένων, η Επιτροπή έχει μειώσει τις φιλοδοξίες της, στις υπηρεσίες αυτές για να δημιουργήσει μια τομεακή νομοθεσία σε αυτό το τομέα. Όμως, για άλλη μία φορά, ο κανονισμός για τις υπηρεσίες στα λιμάνια δεν αντιμετωπίζει τα πραγματικά ζητήματα των λιμένων. Βεβαίως, οι θαλάσσιες μεταφορές ε, είναι ζωτική σημασίας για να υπάρξει μεγαλύτερη βιωσιμότητα στον τομέα μεταφορών. Εμείς ε, θεωρούμε ότι οι λιμένες θα πρέπει να ενταχθούν σε μια ευρύτερη βιώσιμη πολιτική που να αντιμετωπίζει θέματα περιβάλλοντος και κοινωνικά και να υπάρξει συντονισμός μεταξύ λιμένων έτσι ώστε να μπορέσει να εξωτερικευτεί και ένα ενεχόμενο κόστος. Χρειάζεται διαφάνεια. Δεν μπορούμε να μιλάμε για υπηρεσίες χωρίς να λάβουμε υπόψη τις εισρωές δημοσίου χρήματος για τις υποδομές και τις επιχειρήσεις. Ο κανονισμός αυτός θα μπορούσε να έχει διευκολύνει μερικούς από αυτούς τους στόχους. Φαίνεται όμως ότι επιδιώκει να διασφαλίσει ένα δίκτυο διασύνδεσιμότητας. Ως προς την ε, χρηματοδοτική διαφάνεια δεν γίνονται αρκετά έτσι ώστε να φτάσουμε στη νομική ασφάλεια που επιβάλλεται για τον τομέα, γιατί θα πρέπει να υπάρχει χρηματοοικονομική διαφάνεια και ε, μπλοκάρισμα των ε, κρατικών ενισχύσεων και οι δύο προτάσεις θα έπρεπε να είχαν ε, προωθηθεί παράλληλα. Όταν ε, μιλήσαμε για αυτή την πρωτοβουλία 11 χρόνια πριν, η Επιτροπή ήθελε να ορίσει κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές επιδοτήσεις πριν από το 2017. Είναι πολύ απογοητευτικό, αλλά δεν μας εκπλήσει. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεχτεί αυτή την έκθεση, θα πρέπει να δεχτεί σοβαρές επικρίσεις, διότι πρόκειται για μία νομική δέσμευση η οποία δεν κάνει τίποτα για την πραγματική αντιμετώπιση του ζητήματος. Αυτή η νομοθεσία είναι αναποτελεσματική και γι' αυτό θα ήθελα να απορρίψετε αυτή την έκθεση όταν ψηφίσετε αύριο. Ευχαριστώ. Κύριε Τέιλορ, δέχεστε ε, μία μπλε κάρτα από την κυρία Κίρτον Ντάρλιν. Ευχαριστώ κύριε Τέιλορ. Συμφωνείτε ότι αυτό το πακέτο, αν και είναι βελτιωμένο, ενέχει τους ίδιους κινδύνους με την πρόταση που είχαμε απορρίψει το 2006 με μεγάλη πλειοψηφία. Επιβάλλει μεγαλύτερο διοικητικό φόρτο για τα λιμάνια χωρίς να υπάρχει προστασία ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων ή προστασία στην εργασία. Έχετε απόλυτο δίκιο, λέει ο κύριος Τέιλορ, και μην ξεχνάτε ότι το Κοινοβούλιο είχε απορρίψει αυτές τις προτάσεις δύο φορές μέχρι τώρα. Δεν υπάρχουν ε, περιβαλλοντικές απαιτήσεις, γίνεται λόγος για μελέτη αντικτύπου, για, τη, για περιφαλλοντικά ζητήματα, όλα αυτά έχουν διαγραφεί. Δηλαδή προσπαθείτε να προωθήσετε στο Κοινοβούλιο μία νέα εκδοχή του ίδιου πράγματος. Γι' αυτό θα πρέπει να πούμε ανερυθρία στα όχι. Από, το, από την Ευρώπη για τη Δημοκρατία, ε, Jill Seymour για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ο κανονισμός για τις λιμενικέ υπηρεσίε. δεν είναι επιθυμητός στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σε αντίθεση με την Ευρωπαϊκή Υπερό, η Βρετανία έχει πολύ ανταγωνιστικά λιμάνια με τον ιδιωτικό τομέα η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπάθησε να ρυθμίσει το θέμα αυτό ανεπιτυχώς και αυτή είναι η τρίτη προσπάθεια. Καθώς τα περισσότερα λιμάνια στην Μεγάλη Βρετανία είναι ιδιωτικά και πάρα πολύ αποτελεσματικά δεν απόκειται στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ρυθμίσει αυτό το θέμα. Με το δημοψήφισμα για το Brexit ο Βρετανικός λαός ε, θα ψηφίσει την ε, αποχώρηση και θα ε, ανακτήσουμε και πάλι την ελευθερία μας να διαχειριζόμαστε τις δικές μας ε, επιχειρήσεις. Η Μεγάλη Βρετανία έχει μια μακρά προϊστορία όσον αφορά τις εμπορικές σχέσεις με τον υπόλοιπο κόσμο και ο τρόπος αυτός την οδήγησε σε μια μεγάλη ευημερία. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Αρνοτή Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η απελευθέρωση των λιμενικών υπηρεσιών είναι κάτι το παλιό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην αρχή της δεκαετίας του 2000 η Κομισιόν απέτυχε δύο φορές. Επανέρχεται λοιπόν. Η πρόταση της Κομισιόν είναι απαράδεκτη. Αφενός είναι μια απόπειρα ε, να γίνουν ε, ομοιογενή τα λιμάνια που έχουν διαφορετική οργάνωση ε, υποχρεώνοντας τα κράτη-μέλη να στελεχώνουν ε, τα λιμάνια βάσει της πύρας για να προσελκύσουν περισσότερες επενδύσεις βασίζεται στην ανάγκη απελευθέρωσης ορισμένων υπηρεσιών πράγμα που θα εμποδίσει ε, τις, τα κράτη-μέλη να γίνονται ορισμένες υπηρεσίες ε, κάτω από την εθνική ε, σημαία, να χρησιμοποιούνται άτομα τα οποία δεν είναι ειδικευμένα σε πλοία τα οποία έχουν μια σημαία ευκαιρίας είναι κάτι το απαράδεκτο θα είναι ένα ε, κενό πλαίσιο αυτή ε, ο κανονισμός. Γιατί θέλουμε τα λιμάνια μας στρατηγικό στοιχείο της οικονομίας μας να αγοραστούν από ξένους επενδυτές όπως ήταν η περίπτωση του Πειραιά που αγοράστηκε από την Κινέζικη Κόσκο. Θα ψηφίσουμε κατά της πρότασης της Κομισιόν και κατά της πρότασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Μαρινέσκου. Ε, σας συγχαίρω για τα ρουμανικά σας, κύριε Πρόεδρε. Το θέμα ε, συζητείται και υπάρχουν πολύ ζωηρές συζητήσεις διότι υπάρχουν διστάμενες απόψεις. Όμως φτάσαμε σε ένα συμβιβασμό θα δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης, θα αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα των λιμένων. Θα μπορεί ε, κανείς να ορίσει τους δασμούς και τα τέλη, καθώς και τους ε, ναύλους, αβίαστα, έτσι ώστε να υπάρχουν ίσοι όροι πρόσβασης για όλους και να μην υπάρχει άκερη κρατική επιδότηση. Τα κράτη-μέλη θα έχουν την ευελιξία να μην ε, ε, συμπεριλάβουν τα λιμάνια στα περιφερειακά δίκτυα, αν δεν το επιθυμούν. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να βελτιωθεί η ποιότητα των υπηρεσιών. Επειδή ακριβώς υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός, επίγει να αποφασίσουμε Ελπίζω να αρθούν οι, οι διχασμοί που υπάρχουν. Ευχαριστούμε τον κύριο Μαρνέσκου. Και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Ισμαήλ Ερτούγκ για δύο λεπτά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι, αξιότιμη κυρία Επίτροπε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Φλέκενστάιν, για το δύσκολο έργο που επετέλεσε. Γιατί και ίσως δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι εδώ πρόκειται για μια πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από την ε, εποχή του Κάλλας που είχε σαν στόχο τη μία τούρμπο απελευθέρωση σε όλους τους τομείς. Άρα λοιπόν ήταν πολύ δύσκολο ο εισηγητής να βρει εδώ ένα συμβιβασμό και όπως το λέει και η ονομασία ένα συμβασμός δεν είναι κατά 100% αυτό το οποίο επιθυμούν, επιθυμεί ο καθένας. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει κανείς να είναι διατηθειμένος να προβεί σε συμβασμούς. Εάν δούμε τώρα το κείμενο αυτό στο τραπέζι βλέπουμε ότι η υποχρεωτική απελευθέρωση η οποία ήταν, προβλεπόταν ε, στην αρχή από, ε, από την Επιτροπή ε, έχει αποφευχθεί αυτό το οποίο για μένα ήταν το βασικό επιχείρημα ε, για να το υπερψηφίσω είναι οι λεγόμενες ελάχιστες ε, προδιαγραφές που μπόρεσε να διαπραγματευτεί ο εισηγητής όσον αφορά για παράδειγμα την αναγνώριση ε, της, το θέμα της καλής φήμης όταν δεν τηρούνται οι κοινωνικές προδιαγραφές. Και πραγματικά αυτό είναι ένα όφελος γιατί σε, πολλές, σε πολλά άλλα θέματα δεν ε, πετύχαμε να περάσουμε κοινωνικές ε, πτυχές. Και όσον αφορά το θέμα της ε, διαφάνειας, θεωρώ ότι μπορούμε να συνοψίσουμε όλα αυτά τα πλονεκτήματα και να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι το ποτήρι είναι κατά το ίμιση γεμάτο και όχι άδειο, άρα να, το, να την έκθεση. Τώρα η κυρία Φώστερ έχει το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ειλικρινά τον κύριο Φλέκενστάιν για την σκληρή επίμονη δουλειά πάνω σε αυτό το θέμα. Αλλά δεν πιστεύω ότι οι αλλαγές αυτές ε, προχωρούν αρκετά. Όταν άρχισε η διαδικασία ε, ιδιωτικοποίηση των λιμένων στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, ήταν κάτι, πολύ, κάτι που επέφερε επιτυχία στην οικονομία και στην απασχόληση. Δεν θα κάνω τίποτα το οποίο θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά αυτήν την κατάσταση. Η ε, συντηρητική Πολωνία, αν ε, πιστεύουμε ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ των λιμένων και όχι οι δεσμευτικές διατάξεις είναι καλύτερος ε, κινητήρας για αποτελεσματικότητα. Είναι πολύ γραφειοκρατική πρόταση Κομισιό και δεν ταιριάζει με την οικονομία μας των ιδιωτικοποιημένων υπηρεσιών. Ξέρω ότι τα συνδικάτα και οι ιδιοκτήτες των λιμένων είναι αντίθετοι προς την πρόταση ως έχει. Αυτό το κείμενο θα είναι σαν να επηρεάζονται και να ε, επιβάλλεται στους ιδιωτικούς λιμένες υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας, δημοσίου συμφέροντος. Οι κοινωνικές διατάξεις του εισηγητή ε, και άλλες σχετικά με την μεταφορά προσωπικού όσον αφορά την ε, αλλαγή παρόχου είναι κάτι το οποίο δεν μας κάνει. Είμαστε απογοητευμένοι ότι δεν περιλαμβάνονται οι μικροί λιμένες και για τους λόγους αυτές ε, έχω καταθέσει ε, τροπολογίες που θα εξαιρέσουν τους μικρές λιμένες για να επιτρέψουν καλύτερο ανταγωνισμό και να μπορούν οι λιμένες να παρέχουν καλές υπηρεσίες σε καλές τιμένες. Και επίσης θα πρέπει οι ιδιωτικοί λιμένες να εξαιρούνται. Θα ήθελα ε, ε, να, η προτίμησή μου να είναι να απορρίψουμε την πρόταση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, αγαπητοί συνάδελφοι, ορισμένοι συνάδελφοι δεν είναι απολύτως ικανοποιημένοι, είπαν. Ούτε εγώ, άλλωστε. Το θέμα είναι ποιες είναι οι άλλες εναλλακτικέ λύσεις που έχουμε. Ε, αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι χρειαζόμαστε μια καλύτερη πρόσβαση στις λιμένες, χρειαζόμαστε μια καλύτερη διαχείριση των λιμένων, χρειαζόμαστε μια καλύτερη οργάνωση. Αυτό είναι προφανές. Το θέμα είναι κατά πόσο θα έπρεπε να ζητήσουμε από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς να πετήσουμε να παραμείνουν σε ένα καθεστώς νομικής αβεβαιότητας. Παρόλο λοιπόν που δεν είμαι απολύτως ικανοποιημένος με την πρόταση, θεωρώ ότι έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου να υποβάλουμε κάποιες προτάσεις για τη διαπραγμάτευση. Ε, αυτός γι' αυτό είμαι ε, υπέρ ε, της πρότασης. Κύριε Ταλίτσκα, δέχεστε μπλε κάρτα από την κυρία Μάισνερ. Κυρία Μάισνερ έφερα το συνάδελφο σε δύσκολη θέση γιατί ετοιμαζόταν να φύγει. Αγαπητέ κύριε Τέλετσκα, ναι μεν κερδίσαμε πέντε δευτερόλεπτα, παρόλα αυτά έχω το ερώτημα. Ε, πολλοί είπαν ότι υπάρχει ελάχιστη διαφάνεια και μικρή ευελιξία για τις χώρες μέλη. Επίσης δεν ελήφθη υπόψη το γεγονός ότι οι λιμένες διαφέρουν μεταξύ τους. Επίσης δεν ε, ελήφθη υπόψη το ζήτημα των ιδιωτικών λιμένων. Πώς το βλέπετε εσείς, υπάρχει πράγματι μικρή διαφάνεια και μικρός βαθμός ευελιξίας, συμφωνείτε με αυτό ή όχι. Η οχι Κύριε Μάσα, θα ήθελα να σας πω ότι παρόλα αυτά εγώ βλέπω εδώ μία βελτίωση. Άρα μπορώ να συμφωνήσω. Το θέμα είναι κατά πόσο όλα αυτά αρκούν. Ε, βεβαίως ε, θα ε, χρήζουν ε, βελτιώσεων. Ωστόσο η πρόοδος σε σχέση με προηγούμενες προτάσεις κατ' δεν είναι αμεληταία και είμαι πρόθυμος να την υποστηρίξω για να προχωρήσουμε σε διαπραγματεύσεις. Uh, uh, Η κυρία Κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το κείμενο αυτό έγινε πολλής λόγος για την εθνική πείρα κάθε χώρας. Θα σας εξηγήσω τι συμβαίνει στη χώρα μου, την Φινλανδία. Οι λιμένες τα τελευταία χρόνια γνώρισαν μια πραγματική επανάσταση εφόσον στην αρχή του 2015 έγιναν ε, ε, ανώνυμες εταιρείες με μετοχές και σύμφωνα με τους κανόνες της αγοράς ε, και διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο. Ο κανονισμός για τον οποίο μιλούμε εδώ περιλαμβάνει απαιτήσει που είναι ήδη στην καθημερινή ζωή των ηθινόντων στους φινλανδικούς λιμένες. Νομίζω ότι είναι σημαντικό ούτως ώστε παντού στην Ευρώπη να υπάρχει το ίδιο νομικό πλαίσιο για τις λιμενικές υπηρεσίες και την οικονομική διαφάνεια κυρίως για τις δημόσιες επενδύσεις. Το τελικό κείμενο ίσως δεν είναι τέλειο, αλλά για μένα είναι αρκετά ικανοποιητικό. Ευχαριστώ τον εισηγητή και τους σκιώδεις εισηγητές για την επιμονή τους στην εργασία τους και ελπίζω ότι το κοινοβούλιο μας θα υπάρξει ψύχρεμη μέχρι τέλους και θα ψηφίσει καλά αύριο. Ευχαριστώ. Και τώρα η κυρία Ντουπικέτα Μαντέλη, 1,5 λεπτό. Κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι η τρίτη φορά που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιχειρεί να επιβάλλει απελευθέρωση των λιμενικών υπηρεσιών στην Ευρώπη. Άλλαξε ίσως το όνομα, αναφέρεται οργάνωση λιμενικών υπηρεσιών. Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας πρόκειται να ε, μπουν σε ανταγωνισμό ε, οι πιλότοι, τη ρημούλκηση, οι λιμενισμοί, παρόλο που οι καταστάσει είναι διαφορετικές. Αυτό που ισχύει στην Αμβέρσα, στη Ρότερνταμ, που έχουν 20% της μεταφοράς εμπορευμάτων στην Ευρώπη, δεν μπορούν να ισχύσουν για το Αύρα. Και η μελέτη επιπτώσεων δεν λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες των λιμένων. Ακόμα χειρότερο επιβάλλει μια θεώρηση ομοιογενής βάλος της αλήθειας, της ζωής των ανθρώπων, των απαιτήσεων, των περιβαλλοντικών και κοινωνικών. Ο στόχος μας θα πρέπει είναι να προστατεύσουμε τις ακτές και την ασφάλεια στους λιμένες, αλλά να προστατεύσουμε και τους εργαζόμενους. Η βασική απέτηση των λιμένων των ευρωπαϊκών δεν είναι η απελευθέρωση. Ζητούν μια διασάφηση των κανόνων ε, και εδώ και πάρα πολλές χρόνια η Κομισιό έχει κατευθυντήριες γραμμές για τους λιμένες. Ακόμα και ορισμένες εξαιρέσεις επιτεύχθηκαν στις διαπραγματεύσεις. Το κείμενο αυτό δεν έχει αρκετά αναχώματα για, να, για, την προστασία και δεν μπορούμε παρά να ψηφίσουμε κατά του ε, σχεδίου αυτού. Ευχαριστώ πολύ κυρία Και τώρα το λόγο έχει ο κύριο Σαμάτο. Για ένα λεπτό. Η κυρία. Ευχαριστώ. Φαίνεται ότι ο κανονισμός έχει κατανοήσει τις διαφορές ε, μεταξύ ευρωπαϊκών λιμένων. Απλώς αλλάζει το πλαίσιο υπηρεσιών. Υπάρχει μεγαλύτερη διακριτική ευχέρεια για τα κράτη-μέλη. Δεν μπορεί να ισχύσει όμως κάτι τέτοιο για όλα τα λιμάνια, γιατί διαφέρουν άρδιν μεταξύ τους. Θα πρέπει λοιπόν να γίνουν μεν οι λιμένες πιο ανταγωνιστικοί αλλά όχι με οποιοδήποτε κόστος. Θα πρέπει λοιπόν να εμπλουτίσουμε αυτή την πολιτική με μια κοινωνική διάσταση. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε τον ε, ρόλο των κοινωνικών εταίρων και θα πρέπει να καταπολεμήσουμε την ε, προσωρινή εργασία. Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να προωθηθεί η κοινωνική ασφάλεια, ιδιαίτερα για τους ε, μικρούς λιμένες που δεν θα πρέπει να, έχει το ίδιο, δεν θα πρέπει να έχουν το ίδιο διοικητικό άχθος. Ε, ε ευχαριστώ. Ο κύριος Γκράντες Πασκουάλ έχει το λόγο, το λόγο για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε τα λιμάνια ε, έχει διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο για τη δημιουργία των διευρωπαϊκών δικτύων στις μεταφορές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το γνωρίζει πολύ καλά, γι' αυτό ε, είχε καταβάλει δύο προσπάθειες ήδη και αυτή είναι η τρίτη. Μιλάμε για μεγαλύτερο ανταγωνισμό, διαφάνεια, ίση μεταχείριση, κοινωνική ασφάλεια, αποδοτικότητα. Και παρόλα αυτά υπάρχουν πολλές εξαιρέσεις, ένα μη διαφανές πλαίσιο διαχείρισης των λιμένων. Επίσης, τα κράτη-μέλη ε, επιβλέπουν το ολοκαθεστώς. Όπως ξέρετε, οι λιμένες στην Ισπανία είναι δημόσιοι, άρα δεν, μπορούμε, δεν μπορούν να γίνουν διαπραγματεύσεις με ιδιωτικούς φορείς για να ε, οριστούν οι δασμοί και τα τέλη. Θα καταψηφίσουμε αυτή την έκθεση γιατί δεν τηρούν, τηρούνται οι διατάξεις ε, που απαιτούν τα κράτη-μέλη. Πρόκειται για μία τρίτη προσπάθεια. Λέτε ότι θα είναι η μόνη ε, βιώσιμη προσπάθεια. Αλλά κυρία Επίτροπε, δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι δεν θα είναι ε, ε, δυνατό να υπάρξει συμβίωση των διαφόρων τρόπων μεταφοράς με αυτό που προτείνετε εσείς. Ευχαριστούμε πολύ. Ο λόγος είναι στην κυρία Μπονφά. Ευχαριστώ πολύ. Ε, το κείμενο για τις λιμενικές υπηρεσίες ήταν ε, ένα μυθικό πλάσμα για πολύ καιρό, για το οποίο μίλησαν όλοι, αλλά δεν το βλέπαμε ποτέ. Ωστόσο, μετά από πολλού μήνε δουλειά, ο κύριο ε, Φλόκενστάιν, ο εισηγητή από τη Σοσιαλιστική Ομάδα, εκπώνησε ένα κείμενο το οποίο θα ψηφίσουμε αύριο. Είναι καρπό ε, μακρών διαπραγματεύσεων για να καταλήξει σε συμβιβασμού που άλλαξαν ριζικά την ακραία φιλελεύθερη άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εγώ συνεργάστηκα εδώ και χάρηκα για το έργο του εισηγητού. Ε, πρόκειται για ευαίσθητες υπηρεσίες και θα σταθεροποιηθεί η οικονομικό καθεστώς των λιμένων οι νομικές υποχρεώσεις είναι πολύ ξεκάθαρες ε, στην έκθεση και αυτό οδηγεί σε μια πιο κοινωνική Ευρώπη. Η διαφάνεια επίσης είναι καθοριστικό στοιχείο της έκθεσης και θα επιτρέψει έναν πιο υγιή ανταγωνισμό εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά τα πιο τροτά, οι πιο τροτοί λιμένες δεν θα έχουν υπερβολικό διοικητικό φόρτο. Το κείμενο παρέχει αναγκαίες, αναγκαία κοινωνικά χέγγια, ούτως ώστε να έχουν οι χώρες μέλη ένα αρκετό περιθώριο ελιγμών γιατί πράγματι επικύλουν πάρα πολύ τα μοντέλα οργάνωσης των λιμένων στην Ευρώπη και δεν είναι δυνατόν να επιβάλλουμε με τη δύναμη ένα ενιαίο μοντέλο. Το παρόν κείμενο είναι ικανοποιητικό, δεν θα πρέπει να υπονομευτεί στο πλαίσιο του, της τριμερούς ε, συνάντησης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να φτάσει στη διαπραγμάτευση με την πιο ισχυρή θέση και αυτό θα περάσει μέσα από μια ομοφωνία στην ψηφοφορία. Ε, θα πρέπει λοιπόν να υπερψηφιστεί το κείμενο, ε, το οποίο είναι καλό. Και αυτή τη στιγμή βρεθεί μια ε, συμφωνία με το Συμβούλιο και την Επιτροπή, τότε το Κοινοβούλιο θα μπορέσει να απορρίψει ένα κακό κείμενο. Η κυρία Παραντίκα. Ε, η ανταγωνιστικότητα των λιμένων έχει θέση κλειδί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιθυμούμε να υπάρχει μια αυτονομία στη διαχείριση αυτών των λιμώνων που να ενισχύει τον ανταγωνισμό και τους ίσους όρους για όλους, καθώς και μια μείωση ε, στην γραφειοκρατία, ε, προστατεύοντας ταυτόχρονα τα δικαιώματα των εργαζόμενων με την εγγύηση... Παρακαλώ λίγο βραθύτερα. Ε, ελπίζουμε ότι η αυτονομία των ε, λιμένων, η οποία εκφράζει σε διάφορα διαφορετικά μοντέλα, καθώς και ο, ε, η άξιση του αγωνισμού θα επιτρέψει καλύτερη λειτουργία οι λιμένες ε, χωρίς ε, να χάσουν τον ε, δημόσιο χαρακτήρα τους θα πρέπει να έχουν την διακριτική ευχέρεια να καθορίζουν το ύψος των τελών. Αλλιώς θα υπονομευθεί η αυτονομία τους και η δυνατότητα αυτόνομης διαχείριση των λιμένων. Κυρία Πένιας, για ένα λεπτό. Θα ήθελα να αναφέρω ένα στοιχείο που για μας είναι σημαντικό. Το κέντρο βάρους μεταφέρθηκε από την φιλελευθεροποίηση στο κοινωνικό σκέλος. Δηλαδή μιλάμε για ιδιωτικοποίηση των ε, λιμένων και δυστυχώς καταδικάζεται το κοινωνικό μοντέλο γιατί δεν θα μπορέσουν να, να υπάρξουν καλές υπηρεσίες. Μιλάμε για επιβολή του, της θέλησης των μεγάλων επιχειρήσεων και αυτό οδηγεί σε υψηλότερο κοινωνικό ντάμπινγκ στην Ευρώπη. Αυτό δεν είναι το δικό μας μοντέλο. Θα πρέπει να έχουμε πιο αποδοτικά λιμάνια, βιώσιμα, χωρίς να επιδεινωθούν οι όροι εργασίας και η ποιότητα των υπηρεσιών. Ο κύριος Κόχ για ένα μισή λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, αξιότιμοι συνάδελφοι, μια τάση απελευθέρωσης των λιμενικών ε, υπηρεσιών έχουν υπάρξει και στο παρελθόν το 2001 και το 2004. Τώρα έχουμε ένα τρίτο πακέτο για τους ε, λιμένες. Ήδη από το 2013 γίνεται αυτή η προσπάθεια. Και παρόλο που η σύνθεση του Κοινοβουλίου έχει αλλάξει ριζικά έκτοτε, παρόλα αυτά το σώμα παρέμεινε πιστό στις ε, υψηλές του αξιώσεις ε, η σημερινή έκθεση δεν ε, επιβάλλει την υποχρέωση της ιδιωτικοποίησης. Γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, ο οποίος δεν έχασε το στόχο από τα μάτια του και συνέχισε να αγωνίζεται για την ελευθερία της ε, διοργάνωσης των λιμένων για την κάθε χώρα μέλος. Ε, Βεβαίω ήταν δύσκολο να υπάρξει ένα κείμενο με συνοχή και συνέπεια. Παρ' όλα αυτά θεωρώ το κατάφερο ο εισηγητής και κυρίως χαιρετίζω το ξεκάθαρο αίτημα διαφάνειας επειδή τόσο οι πάροχοι όσο ε, όσον αφορά τόσο τον αριθμό των παρόχων όσο τα τέλη και τα αποτελέσματα για τους ε, χρήστες. Ε, επίσης ε, χαιρετίζω το, συμφωνώ με το θέμα μιας ε, επαρκούς κατάρτισης για τους εργαζόμενους στις λιμενικές υπηρεσίες. Γι' αυτό θα υπερψηφίσω την έκθεση. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό η κυρία Βερμέχο. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να βελτιστοποιήσουμε τους όρους εργασίας των εργαζομένων στα λιμάνια, να μην υπάρξει πλήρης απελευθέρωση θα πρέπει λοιπόν να ορίσουμε νέα, νέες κοινωνικές προδιαγραφές. Θα πρέπει να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας στα λιμάνια. Αυτό το ζητούσαμε ήδη εδώ και πολύ καιρό στον κανονισμό για την απασχόληση. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και συμβάσεις και θα ήθελα να τονίσω ότι αυτό θα πρέπει να ισχύσει και στα δημόσια και στα ιδιωτικά λιμάνια. Δεν δεχόμαστε τις εξαιρέσεις που θέλει η δεξιά. Δεν μπορούμε να έχουμε ανεπαρκή προστασία των εργαζομένων και να μην υπάρχει δημόσια χρηματοδότηση των λιμένων. Δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε την ανάγκη της ε, του δημόσιου ελέγχου των λιμένων. Ο κύριος Σαλίν για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ να σας συγχαρώ για την εξαιρετική εργασία, να ευχαριστήσω και τους ε, και την κυρία Βόζεμπερκ που ήταν σκιώδης από τη δική μου ομάδα. Προσπαθήσαμε να συγκλίνουμε τις ε, διάφορες απαιτήσεις των ε, ευρωπαϊκών λιμένων. Βεβαίως η απάντηση δεν είναι πάντα ικανοποιητική. Όμως κατά τη, βάση, κατά τη φάση της διαπραγμάτευσης και των τριμερών θα προσπαθήσουμε να εγγυηθούμε τα βασικά σημεία όπως είπαμε, τα λιμάνια δεν είναι όλα ίδια. Υπάρχει διαφοροποίηση και διαφορά του τι συμβαίνει στα λιμάνια του Βορρά ή του Νότου. Στην Ιταλία έχουμε ένα μεγάλο μακρύ κατάλογο επιβατών που ε, δαπανούν 7, ε, μάλλον καλύπτουν 7 έως 8 εκατομμύρια ετησίως και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και τα εμπορεύματα αποτελούν το 37% της εσωτερικής αγοράς. Άρα ξέρουμε ότι θα πρέπει να συγκλίνουν όλες οι απαιτήσει. Από αυτή την άποψη και στον κοινωνικό τομέα θα πρέπει να προσέξουμε θα πρέπει τα λιμάνια να είναι τα σημεία όπου συγκλίνουν οι μεγάλες επενδύσεις της Ευρώπης. Ναι στην διαπραγμάτευση, ναι στην έκθεση, αλλά θα πρέπει αυτές οι διαφορετικές απαιτήσεις να συγκλίνουν προς ένα κοινό παρονομαστή. Ο κύριος Φερέιρα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Η εργασία στους λιμένες, η υφίσταται την πίεση των καπιταλιστικών δυνάμεων. Οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι πολυεθνικές θέλουν να συμπιέσουν το κόστος. Γι' αυτό υπάρχει απορρίθμιση και απελευθέρωση των ε, αγορών και των λιμένων κατά συνέπεια. Η κατάσταση στην ε, Πορτογαλία είναι ενδεικτική. Με βάση τον παρεμβατισμό της Τρόικας ε, έγινε μία απαράμιλη εκμετάλλευση και των λιμανιών και θέλετε να προχωρήσετε ακόμα περισσότερο στην εκμετάλλευση. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι ότι υπάρχει μεγάλη μαχητικότητα από τους εργαζόμενους και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να προωθήσουμε τα εθνικά μας συμφέροντα. Κασιεύσκα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το σχέδιο κειμένου ήταν καλύτερο από τα δύο που απορρίφθηκαν στο παρελθόν. Νομίζω ότι μετά από 15 χρόνια η Ευρώπη αξίζει να έχει κανόνες ποιότητας που να μην ε, έχουν ασάφειες και και στον εισηγητή μπορούμε να πούμε ότι η Πολωνία δεν έχει πρόβλημα ε, διαφάνειας. Η Πολωνία έχει κείμενα τα οποία δεν λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των ευρωπαϊκών λιμένων. Ξεκινάμε από την αρχή ότι έχουμε μια μοναδική θεώρηση ευρωπαϊκή που είναι καλύτερη από τις μονομερείς δράσεις των κρατών μελών. Αλλά δεν συμφωνούμε με, ορισμένα πράγματα, με τη γραφειοκρατία με τις αλλαγές στους θεσμούς. Στην Πολωνία έχουμε πολύ καλούς κανόνες που εγγυώνται την οικονομική διαφάνεια, την οικονομική ελευθερία, τον ανταγωνισμό, την απαραίτητη παρακολούθηση. Αναπτύσσονται πολύ καλά οι λιμένες στην Πολωνία και φοβούμαστε μήπως οι διατάξεις αυτές θα ε, θέσουν σε κίνδυνο την καλή ανάπτυξη. Γι' αυτό η αντιπροσωπεία της Πολωνίας θα ψηφίσει κατά του κειμένου αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα περνάμε στην διαδικασία Catch the Eye. Έχουμε πάρα πολλές αιτήσεις. Αρχίζω με τον κύριο Πούλτσακ. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα να εκφράσω την ελπίδα μου ότι αυτή η τρίτη απόπειρα τελικά ε, θα ευοδοθεί. Χαιρετίζω το γεγονός ότι κατά κάποιο τρόπο αποσύραμε ορισμένα ε, μέτρα ε, του κοινωνικού κεφαλαίου. Αλλά αυτό που είναι σημαντικό είναι η Κομισιόν προωθήσει πραγματικά εναρμονισμένους κανόνες για τους φορείς των λιμένων, ούτως ώστε να υπάρξει αρκετός ανταγωνισμός, διότι έχουμε πάρα πολλές καταχρήσεις καταστάσεων στην αγορά, ε, όσον αφορά κυρίως τις υπηρεσίες διέλευσης, παρόλο ε, που εμείς η τσεχική δημοκρατία δεν έχουμε πρόσβαση στη θάλασσα. Θέλουμε να υπάρχει πλήρης ανταγωνισμός. Ο κύριος Χόουιτ έχει το λόγο. Εδώ ε, ε, οι λιμένες που αντιπροσωπεύω είναι κινητήρας ανάπτυξης και έχουμε το μεγαλύτερο λιμένα ε, εμπορευματίων πύλη προς ε, την Ευρώπη και έχουμε επίσης τις διάφορες ε, υπηρεσίες που παρέχονται που είναι σημαντικές. Έχουμε επίσης σημαντικά στοιχεία για την οικονομία. Ο φίλος μου, ο Φίλκενστάιν, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τις διαπραγματεύσεις για να ενθαρρύνει τον ανταγωνισμό μεταξύ των ευρωπαϊκών λιμένων και ίσους όρους ε, μεταξύ των ε, λιμένων. Επίσης ε, θα πρέπει οι ενώσεις για την ρημούλκηση να έχουν μέτρα για να προληφθεί κάθε καταστροφή θα πρέπει να προσπίσουμε της 146-147 της τροπολογίας για να ενισχύσουμε την διαπραγματευτική ικανότητα. Θα πρέπει να προωθήσουμε την απασχόληση της ε, επενδύσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Χόουιτ. Η κυρία Τόμασιτς. Η έκθεση αυτή τροποποιεί την αρχική πρόταση της Κομισιόν ε, χαίρομαι που δεν θα υπάρχει ενιαίο σύστημα διαχείρισης γιατί θα πρέπει να δεχτούμε την ποικιλότητα των, και την διαφορετικότητα των ε, λιμένων μας. Χαίρομαι ε, γιατί λάβατε υπόψη αυτή τη διαφορετικότητα καθώς και τα, τις σκηνές ελάχιστες προδιαγραφές. Πολύ Συχνά προσπαθούμε να βρούμε καθολικές λύσεις, όμως η έκθεση αυτή αποτελεί εξαίρεση και θα πρέπει να την υποστηρίξουμε. Μιλάμε για χρηματοοικονομική διαφάνεια ως προς την αρχή της αναλογικότητας έχει μεγάλη σημασία διότι τα τέλη δεν θα είναι ασύμφωνα και αυτό είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Αγαπητοί presidenta Αγαπητή Επίτροπε Μπούλτς, αυτή η προσπάθεια θα ορίσει ένα ίσο ε, επίπεδο πρόσβασης και θα προωθήσει και την ανταγωνιστικότητα. Μέχρι τώρα υπήρχε ένας πολύ συγκεντρωτικός χαρακτήρας διαχείρισης χωρίς να λάβουμε υπόψη τους καταναλωτές και την οικονομική ανάπτυξη. Η Ευρώπη θα πρέπει να ακολουθήσει τις ε, χρηστές πρακτικές όπως και την ε, φορολογική αυτονομία. Ως Καταλανός δέχομαι αυτή την έκθεση και ελπίζω να τα καταφέρουμε με ελάχιστες αλλαγές μετά τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Σόλτες. Σόλτες. E, Κυρία αυτός ο κανονισμός ε, σύμφωνα με τους ε, συντάκτες του θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητα και θα μειώσει την γραφοκρατία και σύμφωνα με την Επίτροπο εξεχρονίζει τους λιμένες και μας τρέφει προς το μέλλον. Ε, φυσικά οι λιμένες αποτελούν μια πύλη προς τον κόσμο και έχει λεχθεί ότι το θέμα αυτό συνδέεται με το ζήτημα της απασχόλησης. Όλοι επιθυμούμε αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας με ικανοποιητικές αποδοχές. Όλοι ελπίζουμε επίσης να συνεχίσουν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις με έναν ορθό τρόπο. Γι' αυτό είμαστε υπέρ της ε, υπέρ της ασφάλειας και υπέρ των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Επιθυμούμε επίσης ισότιμους όρους και σε σχέση με τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναμένω να, το, να μεριμνήσει γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση και να μεριμνήσει επίσης και για μια ισορροπημένη ανάπτυξη των λιμένων. Ο κύριος ε, Χέκε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε πάρα πολλές ε, θέσεις εργασίας ε, στους λιμένες και θα εξαρτηθούν οι θέσεις αυτές από την επιτυχία των λιμένων. Δεν πρέπει να έχουμε περισσότερες ρυθμίσεις ε, ενώ έχουμε το εμπόριο με τον υπόλοιπο κόσμο. Θα έχουμε και το δημοψήφισμα γιατί να επηρεαστεί το εμπόριο που δεν έχει να κάνει τίποτα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό είμαστε αντίθετοι για αυτούς τους λόγους. Οι καλύτεροι για να διαχειρίζονται ε, τους ελιμένες μας είναι ο ίδιος ο Βρετανικός λαός. Κυρία Μπατ, Μπάλκ. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να μιλήσω εκ μέρους της Βορείου Ιρλανδίας που θα απογοητευτεί από αυτές τις προτάσεις. Είναι ένα άλλο παράδειγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θέλει να επιβάλλει μια ενιαία λύση, μια λύση που να κάνει για όλους ενώ εμείς έχουμε ε, ανταγωνιστικές συνθήκες. Έχουμε στο Belfast 700 εταιρείες που βρίσκονται στο λιμένα και 2.000 ε, άτομα απασχολούνται εκεί. Έχουμε ε, χίλιες ε, θέσεις εργασίας με μισθούς 26 εκατομμυρίων στην τοπική οικονομία. Δεν θα πρέπει να θέσουμε σε κίνδυνο τα πλεονεκτήματα αυτά για τον τοπικό πληθυσμό. Δεν θέλουμε να έχουμε γραφειοκρατικά εμπόδια. Αν έχουμε υπερβολικές ρυθμίσεις και εποπτεία που ε, θα τιμωρούν ε, τους παρόχους λιμενικών υπηρεσιών. Και αυτό θα είναι μόνο η αρχή. Ε, αύριο θα ψηφίσω κατά της κανονισμού αυτού για να προστατεύσω την οικονομία της Βόρειας Ιρλανδίας. Υπάρχει μια μπλε κάρτα. Κύριε Φλίκενστάιν, έχετε. Δέχεστε την μπλε κάρτα. Ναι, ναι, ναι, για σας είναι. Ναι. Εν συντομία, κυρία συνάδελφε, μπορείτε να μου αναφέρετε δύο ή τρία παραδείγματα τι εννοείτε όταν, όταν θέλετε να προστατεύσετε την οικονομία της ε, Βόρειας Ιρλανδίας. Τι είναι αυτό που την ε, απειλεί συγκεκριμένα. Γιατί πιστεύω ότι οι λιμένες της ε, Βορείου Ιρλανδίας μπορούν να επωφεληθούν τα μάλα γιατί δεν είναι καθόλου υποχρεωμένοι να αλλάξουν τίποτα εδώ. Ευχαριστώ τον εισηγητή για την ερώτησή του. Θα ήθελα να επιβεβαιώσω ότι ήρθα σε διαβούλευση με τα λιμάνια της Ιρλανδίας της Βόρειας Ιρλανδίας που αντιτίθενται σε αυτές τις αλλαγές θεωρούν ότι πλήττουν τον, την ανταγωνιστικότητα και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Και σε αντίθεση με, το, με άλλες πόλεις, το Belfast έχει μεγάλη σημασία οι 22.000 θέσεις οι οποίες ε, τώρα ε, τίθενται εν κινδύνο. Κέλλη. Όπως ξέρετε, επειδή προέρχομαι από την Ιρλανδία, τα λιμάνια έχουν μεγάλη σημασία για μας. Νομίζω ότι αν λάβουμε υπόψη και τα μελλοντικά χρόνια θα υπάρξουν μεγάλες αλλαγές στις θαλάσσιες μεταφορές. αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρχει διαφάνεια, σωστός ανταγωνισμός και ε, ασφάλεια εργασίας. Γι' αυτό θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα στο Σάνον, στη δική μου ε, εκλογική περιφέρεια. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η διόρυγα του Παναμά Τώρα έχει διπλασιάσει τη χωρητικότητά της, οπότε καταλαβαίνει τι ανταγωνιστικότητα υπάρχει έναντι της Ευρώπης, κάτι το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι η τρίτη προσπάθεια και εδώ για τους λεμένες και θα ήθελα να δούμε τι σημαίνει ο Επίτροπος κύριος Γάλλας ήθελε να εφαρμόσει κανόνες ανταγωνισμού εντός των ε, λιμένων επιβάλλοντας μια δυναμική ανταγωνισμού ε, σε όλους τους ε, λιμένες. Αλλά επιθυμώντας επίσης να κατοχυρώσουν την ασφάλεια των εργαζομένων. Για τα για τα λιμάνια της Νότιας Ευρώπης είναι μια ευκαιρία να δημιουργηθούν συνθήκες ασφάλειας και σε σχέση με τα λιμάνια της ε, Βόρειας Ευρώπης τα οποία έχουν πολύ περισσότερες ε, ενισχύσεις. Η κυρία Πέτροπος ε, έθεσε το θέμα της ενίσχυσης των υποδομών των λιμένων. ευχαριστώ κυρία πρόεδρε η πρόταση είναι καλή όντως καθυστέρησε ε, δεν είναι τέλεια αλλά σε τελική ανάλυση υπάρχουν περισσότερα στοιχεία θετικά παρά αρνητικά. Οι ευρωπαϊκοί λιμένες χρειάζονται δίκαιους κανόνες που δεν θα αποκλείουν κανέναν, χρειάζεται διαφάνεια για το καλό όλων. Αυτή η πρόταση, κατά τη γνώμη μου, ενισχύει όλα αυτά τα στοιχεία και για τον λόγο αυτό την υποστηρίζω. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπούλτσο έχει τον λόγο. Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Άκουσα με μεγάλη προσοχή τα σχόλια όλων σας, αλλά ορισμένες πληροφορίες ε, ίσως είναι κάπως απαρχαιωμένες, διότι οι εξαιρέσεις ε, για τις κρατικές επιδοτήσεις δημοσιεύτηκαν σήμερα. Και αυτό που έχει σημασία είναι τα λιμάνια να γίνουν πιο πράσινα πιο καινοτόμα και ε, γενικότερα να υπάρχει βιωσιμότητα. Αυτό που έχει σημασία είναι να λάβετε υπόψη ότι το κείμενο βασίζεται σε συμπληρωματικά μέτρα εθνικού και κοινοτικού χαρακτήρα έτσι ώστε να μπορέσουν και οι τοπικές αρχές να παρέμβουν. Όπως σας είπα, η δική σας ψήφος θα είναι αποφασιστική σημασίας για να οριστεί ένα νομοθετικό πλαίσιο για τα λιμάνια, έτσι ώστε να ε, λειτουργήσει πολύ σωστά το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών και να φτάσουμε και σε νέες δυνατότητες απασχόλησης. Σε σχέση με ορισμένα από τα σχόλιά σας, οι Άντερσον Γκράντες και Αγιάλα Σέντερ μίλησαν ε, για το θέμα της αυτονομίας των λιμένων θα συνεργαστώ μαζί σας επικοδομητικά στους τριμερείς διαλόγους. Όπως και το Συμβούλιο, πολλοί πιστεύετε ότι ο κανονισμός δεν θα επιτρέψει στα κράτη-μέλη να έχουν λόγο. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Η Επιτροπή θα ε, συζητήσει αυτό το ζήτημα κατά τους τριμερείς. Κυρία Φώστερ, σε σχέση με τα ιδιωτικά λιμάνια, ε, θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν καταχρήσεις δεσπόζουσας θέσης και στρέβλωση του ανταγωνισμού με άλλα λιμάνια. Προς τους Τέιλορ, Ντέιλι και Σόλτες θα ήθελα να σας πω ότι θα πρέπει να υπάρχει ε, outsourcing για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στα τέλη στα λιμάνια και να υπάρξει χρηματοοικονομική διαφάνεια για την πρόσβαση στην αγορά έτσι ώστε να ενθαρρύνουμε τις επενδύσεις για να γίνουν πιο πράσινα τα λιμάνια. Δεν βλέπω να υπάρχει ε, κάποια διαφωνία εδώ με, τις, με τους στόχους, εκπεφρασμένους στόχους των πρασίνων σε σχέση με το άρθρο 10 για τη μεταφορά δικαιωμάτων. Θα ήθελα να είμαι ξεκάθαρη. Δεν θα πρέπει να ρυθμιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτό το ζήτημα. Είναι θέμα εθνική αρμοδιότητας και θα πρέπει να σεβαστούμε το εθνικό εργατικό δίκαιο καθώς και τις ρυθμίσεις στις οποίες έχουν καταλήξει οι κοινωνικοί εταίροι. Είμαι πεπισμένη ότι θα μπορέσουμε κατά τη διάρκεια του ημερούς διαλόγου να ε, επιβεβαιώσουμε και αυτά τα ζητήματα. Ελπίζω έτσι να κάλυψα την ε, κυρία Άντερσον. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή και τους ε, σκιώδεις ε, για την επιμονή που δείξανε. Η υποστήριξη από όλους τους βασικούς φορείς δείχνει ότι είναι ισόρροπη η πρόταση που έχουμε επιτάπητος και έτσι είναι μεγάλες οι πιθανότητες ε, στο μέλλον ε, να επιτύχουμε το στόχο μας ε, με την κατάλληλη στηρίξη ούτως ώστε να έχουμε μια σύρροπη συμφωνία για τους λιμένες, μια συμφωνία που θα ενισχύσει περαιτέρω την ενιαία αγορά και τον ενίο χώρο μεταφορών ένα, από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ζητώ την υποστήριξή σας. Πιστεύω ότι είμαστε έτοιμοι για τριμερείς διαλόγους που θα μας οδηγήσουν στην ε, τελική λύση. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Φλέκενστάιν. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, υπήρξε μακρά και σε βάθος συζήτηση κυρίως με τις λιμενικές αρχές, ε, τις αρχές για τα terminals και τα συνδικάτα. Επί τόπου στο ε, Μπιρεά, στη Ριέκα, στο Κόπερ, στην Βαρκελόνη και στο Αμβούργο. Γνωρίζαμε ότι μετά από την ολέθρια προϊστορία του πακέτου για τα λιμενικά, μόνο τότε μπορεί να υπάρξει συμβιβασμός όταν οι περισσότεροι εμπλεκόμενοι θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Μετά από 15 ε, χρόνια συζητήσεων και αντιπαραθέσεων και μετά από ε, ε, επιθέσεις που είχαν υποστεί και τα κτίρια και στο Στρασβούργο, μετά από πολλή δουλειά υπάρχει η επίτευξη αυτού του στόχου ολοκληρώνοντας θέλω να σας διαβάσω από ένα μήνυμα ηλεκτρονικό που πήρα πριν από κάποιες μέρες. Στις 8 Μαρτίου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ψηφίσει την έκθεση Φλέκενστάιν για την πρόταση για την ρύθμιση των λιμένων. Οι ευρωπαϊκές οργανώσεις που εκπροσωπούν τους λιμένες εκτιμούν τις προσπάθειες που επενδύθηκαν και έγιναν από τον εισηγητή και του γεώδεις εισηγητές για να επιτευχθεί ένα ισορροπημένο κείμενο συμβιβασμού ώστε να ολοκληρωθεί ο διάλογος με τους εμπλεκόμενους. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η εργασία που επετεύχθη μέχρι σήμερα, το έργο που επετεύχθη από τον εισηγητή και τους κοιόδης πρέπει να υποστηριχθεί από την Ολομέλεια και είναι μια πάγια στεναρή βάση για τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Αυτό από πλευρά της Γενικής Γραμματέως της ΕΣΠΟ των ΦΡΙΠΟΣ, των ε, της γραμματείας των ε, ε, θεμάτων αλληλείας και λιμένων και από τον Γενικό Γραμματέα των Υπεύθυνων Λιμενικών Θεμάτων και των Πλοιάρχων και η ερώτηση προς τους επικριτές είναι μήπως θα μπορούσε να υποτεθεί ότι όλοι εκείνοι που θα εργαστούν στο μέλλον με αυτά τα θέματα και συνιστούν να υπερψηφιστεί αυτό το πακέτο μέτρων μήπως δεν κάνουν λάθος όλοι αυτοί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ολοκληρώνω τη συζήτηση. Αύριο θα γίνει ψηφοφορία για αυτή την έκθεση. Ε, θα διακόψουμε μόνο δύο λεπτά για να έρθει στο έδρανο η κυρία ε, Γεωργίευα. Ευχαριστώ. Βάσει τη μεσής διάταξη ε, εξετάζουμε την ετήσια έκθεση 2014 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων τη Ευρωπαϊκή Ένωση κατά πολέμηση απάτη. Ε,